morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dear colleagues, if you may take your seats. Καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν έχω άλλες ανακοινώσεις, εκτός από το να σας ανακοινώσω ότι λόγω της ε, απεργίας που λαμβάνει η χώρα, των ε, κινητοποιήσεων που λαμβάνει η χώρα στις Βρυξέλλες, δεν θα σερβιριστεί καφές, οπότε θα πρέπει εσείς μόνοι σας να σερβιριστείτε από το αυτοσχέδιο καφενείο που βρίσκεται στο πίσω μέρος της αίθουσας. Είναι το καφενείο εκστρατείας της Επιτροπής μας. Σας υπενθυμίζω επίσης. Ψηφίζουμε. Θυμηθείτε τις κάρτες σας. Ερχόμαστε στο σημείο 16. Κατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων. Η εισηγήτρια η κυρία Ναταλή Γκρισπέκ και θα μας παρουσιάσει Θα ακούσουμε τώρα την παρουσίαση του εγγράφου εργασίας της που έχει προετοιμάσει Ακούσαμε για το σχέδιο εφαρμογής από την Κομισιόν και το χρονοδιάγραμμα και η κυρία Γκρίσπακ θα μας παρουσιάσει τα πεπραγμένα της πρώτης συνάντησης των σκιωδών εισηγητών και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση. Κυρία Γκρίσπακ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα το πρωί θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω αυτό το έγγραφο εργασίας, το οποίο έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, για την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ένωση. Αυτό το πρόβλημα είναι κάτι που μας απασχολεί. Έχουμε επίγνωση ε, της έκτακτης ανάγκης ε, και ε, της σημασίας και κάναμε έκθεση πρωτοβουλίας ε, για, κάνουμε προτάσεις γιατί κάθε χρόνο χιλιάδες παιδιά, παιδιά πάση περιπτώσει ανήλικοι, δηλαδή παιδιά και έφηβοι από τρίτες χώρες οι ε, απάτριδες φτάνουν στην Ένωση και είναι εγκατελειμμένοι στη μοίρα τους. Να σας δώσω και μερικά πρακτικά στοιχεία ενημέρωση για το πώς προχωρούν οι εργασίες επ' αυτού επεκτείναμε λίγο, παρατείναμε μάλλον το χρονοδιάγραμμα. Είναι έγγραφο εργασίας στο οποίο θα σας παρακαλούσα συνάδελφοι να μου κάνετε όσο περισσότερες παρατηρήσεις, προτάσεις και κριτικές θέλετε για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια έκθεση έτσι πιο εμπεριστατωμένη και πιο συνεκτική στο τέλος των εργασιών μας. Ε, θα μεταβεί και αντιπροσωπεία αρχές Απριλίου κατά την Τυρκουάς εβδομάδα ακριβώς για αυτό το θέμα της έκθεσής μου ε, και τέλη Απριλίου θα σας κάνουμε την έκθεση. Έχετε λάβει λοιπόν ένα έγγραφο εργασίας που έχει στόχο να βάλει τα θεμέλια, ε, να κάνει προτάσεις. Είμαστε πάρα πολύ ε, ελεύθεροι σε αυτό το θέμα, σε τέτοιου είδους υποθέσεις, για να εντοπίσουμε ε, τα ζητήματα και τα προβλήματα που έχουν σχέση με τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Και επειδή το έχω συζητήσει ήδη με τους κοιόδες ηγητές, θέλω να προσθέσω ότι αυτό το έγγραφο εργασίας δεν είναι ούτε εξαντλητικό, ούτε αποκλειστικό. Επί της ουσίας θα ενταχθεί στο σχέδιο έκθεσης και τις επόμενες εβδομάδες. Ε, θα σας προτείνω να συμπεριλάβουμε όλα τα βασικά ζητήματα, ανησυχίες και θέματα που πρέπει να ε, αναφέρουμε. Ελπίζω οι εβδομάδες αυτές να είναι παραγωγικές, να μπορέσουμε να εργαστούμε ουσιαστικά και ποιοτικά και το κείμενό μας να είναι στο ύψος των περιστάσεων και των αναγκών αυτών των αλληλίκων που ε, είναι και πολύ ευάλωτοι παντού στην Ευρώπη. Για να μπούμε τώρα λίγο σε λεπτομέρειες ε, στο σχέδιο αυτό το έγγραφο εργασίας, τι λέω. Σήμερα, και αυτό πραγματικά κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα θεμελιώδη δικαιώματα των ασυνόδευτων ανηλίκων δεν γίνονται σεβαστά ή γίνονται λίγο σεβαστά σε διάφορα κράτη-μέλη. Ε, ε, υποδοχή, ταυτοποίηση, περίθαλψη, ενασχόληση μαζί τους, πρόληψη ακόμα, είναι ζητήματα ε, και πολλές φορές μεγάλες προκλήσεις και για τα κράτη-μέλη και για την Ευρώπη. Ποια είναι η βασική ιδέα και η κεντρική και νομίζω συμφωνούμε πολύ σε αυτή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προχωρήσει έτσι περαιτέρω για την ε, υποδοχή τους, προστασία τους, ε, για να καλυφθούν όλα τα ελλείμματα και τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των ασυνόδευτων ελίκων. Παρόλο που γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα καθεστώτα που ισχύουν από χώρα σε χώρα προ αυτό. Δύο είναι οι άξονες του εγγράφου εργασίας. Το πρώτο, το ανώτατο συμφέρον του ε, ανηλίκου και μάλιστα το πρόβλημα, βέβαια, όχι πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα, αλλά πρέπει να δούμε πώς ορίζεται αυτό το ανώτερο συμφέρον. πολύ συχνά μας απασχολεί αυτό και το συζητούμε εδώ, θα πρέπει πάντα να κυριαρχεί. Αυτό να είναι το πρώτο μέλημά μας. Πρώτα το παιδί ή ο ανήλικος σε πάση περιπτώσει. Και το δεύτερο είναι αυτό που έχει να κάνει με την προστασία γενικότερα των ανηλίκων. Δηλαδή να μην χρησιμοποιούμε το πρίσμα που συχνά χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη, όχι όλα, πολλά, το βλέπουν αυτό υπό το πρίσμα του ελέγχου της μετανάστευσης. Άλλο αυτό και άλλη προστασία των ανηλίκων. Αυτά τα δύο προτείνω ως ηρμό ε, της έκθεσής μου. Μετά θα πρέπει να λύσουμε πολλά ζητήματα, να απαντήσουμε σε πολλά ερωτήματα, περίπλοκα, ιδιαίτερα. Και τα κράτη-μέλη τα αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο. Τι θέλετε όμως αυτά. Πρώτον, πώς ε, θα ξεπεράσουμε την έλλειψη ή την πλήρη απουσία στατιστικών για ε, τους ασυνόδευτους ανηλίκους στην Ευρώπη. αφορούν διάφορα αριθμητικά στοιχεία. Ερώτηση δεύτερη. Πώς θα χειριστούμε την άφηξη και την ε, ταυτοποίηση. Γιατί και από τη στιγμή που θα ταυτοποιήσει ένα ανήλικο είναι το πρώτο βήμα για την προστασία του. Ποιοι είναι οι κανόνες για την ε, ε, υποδοχή τους και πώς θα δίνεται στους ανηλίκους ουσιαστική πρόσβαση σε ειδικέ υπηρεσίες. Χρειάζονται κοινέ κατευθυντήριες γραμμές για την επιμέλεια τους γιατί διαφέρουν από κράτο σε κράτο, οι αρμοδιότητε, κράτος, τοπική αυτοδιοίκηση και στα ομοσπονδιακά κράτη. Υπάρχει το επίπεδο της κεντρικής κυβέρνηση, η επικεντρωμένη διοίκηση στα κεντρικά, συγκεντρωτικά κράτη κτλ. Και κατά πόσο μπορεί η Ευρώπη να ε, έχει μια κοινή μέθοδο για ε, τον καθαρισμό της ηλικίας. Ε, πώς θα έχει πρόσβαση σε βασικές ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες ε, Λοιπόν, είναι μια σειρά από ερωτήματα για διάφορα κριτήρια, διατρέχουν ε, το έγγραφο εργασίας. Υπάρχει το θέμα του σεβασμού, του ανωτέρου συμφέροντος του ανηλίκου και πώς μπορούμε να προστατεύουμε τα παιδιά αυτά αυτή τη στιγμή ενδεχομένως επαναπατριστούν. Δηλαδή, ποιες είναι οι βιώσιμες λύσεις που μπορούμε να τους προσφέρουμε ε, στους ανηλίκους αυτούς, εάν εγκατασταθούν στην Ένωση, εάν ε, αποχωρήσουν. Και ένα άλλο θέμα που δεν εξετάζεται και δεν αντιμετωπίζεται καλά σε όλες ε, τις περιπτώσεις είναι τι θα γίνει τη στιγμή που θα ενηλικιωθεί ο, ε, ο ανήλικος. Δηλαδή σαν τη σταχτοπούτα από τη στιγμή που πάβει να είναι 17 χρονών και γίνεται 18 η άμαξα ξαναγίνεται κόλο και, θα, και χαιρετίσματα όλα τα υπόλοιπα που γνώριζε όταν ήταν ανήλικος επαναπροωθείται στην πατρίδα του αυτή στιγμή ενηλικιωθεί. Λοιπόν, τα προβλήματα αυτά είναι πάρα πολύ περίπλοκα, πάρα πολύ έντονα και θα άξιζαν πάνω από 4-5 σελίδες που μας επιτρέπουν για τις εκθέσεις πρωτοβουλίας. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα. Θα πρέπει να βρούμε κάποια βασικά, κάποια κόμβικά και να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις εξ στο του Κοινοβουλίου. Προσωπικά θα επιθυμούσα, αλλά περιμένω να ακούσω τι θα πούν και όλοι οι συνάδελφοι, να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάτι που να μας ενώνει και να μας είναι χρήσιμο. Λέω λοιπόν ότι προσωπικά θέλω η έκθεση να είναι πυκνή, συνεκτική, σύντομη, ισχυρή για να μπορέσει να βοηθήσει να αυξηθεί η συνειδητοποίηση για τα ειδικά προβλήματα των ασυνόδευτων αλληλίκων. Γιατί υπάρχουν κείμενα βεβαίως και νομικές βάσεις, αλλά είναι διασκορπισμένα. Έχω και μια ελπίδα, μάλλον φρούδα, να μην έχει μόνο συστάσεις αυτό το έγγραφο για ε, τις ελάχιστες προδιαγραφές, αλλά να είναι και ένα πρακτικό εργαλείο. Φερρυπίν νομοθετικής φύσεως για τα κράτη-μέλη. Και για να ολοκληρώσω θα ήθελα να πω ότι δεν θα πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι ένας ανήλικος πρώτα απ' όλα είναι παιδί. Δηλαδή ένα ευάλωτο ε, πλάσμα ε, και στην Ευρώπη και στα κράτη-μέλη θα πρέπει να το καταλάβουν τα κράτη ε, ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δηλαδή, όχι μόνο να μην ε, ασκείται βία εις βάρος τους, αλλά να προστατεύονται και να λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματά τους. Λοιπόν, ολοκληρώνω για δεύτερη φορά, <laughs> για να περάσουμε στη συζήτηση, Πρόεδρε. Έχουμε όλα τα κείμενα που έχουν σχέση με αυτό στο παράρτημα. Λίγη περίπου το πρόγραμμα δράσης 2010-2014 ε, για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και θα ήθελα να μάθω πώς ε, φρονεί να προχωρήσει στο μέλλον Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υποθέτω ότι θα υπάρξει έκθεση αξιολόγησης, αλλά από εκεί και πέρα τι θα κάνει. Πρόγραμμα δράσης, κάτι πιο δεσμευτικό για να πλησιώσει και συνδέσει και τι δικέ μα εργασίε. Καταλαβαίνουμε ότι η ασυνόδευτοι είναι μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να λυθεί και με χαρά προσβλέπω στη συνεργασία με του συναδέλφου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά μακρηγόρησα λίγο, Πρόεδρε, το ξέρω. Τι να κάνουμε. Ευχαριστούμε, κυρία Γκρισμπέκ. Ανοίγουμε τώρα το, δίνουμε το λόγο τώρα. Και θα ήθελα καταρχά να ρωτήσω του σκιώδεις συζητητές, η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω την Αταλή για το εξαιρετικό της έργο για τη σύνταξη ενός κειμένου που αποτελεί μια θαυμάσια βάση και τονίζει όλα τα σημεία κλειδιά με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούμε. Είναι ένα έγγραφο που παρουσιάζει πολλές προκλήσεις. Βέβαια, πρέπει να είμαστε συνεπείς, σαφείς και περιεκτική. Δεν ξέρω, δεν είμαι βέβαιη. Αυτό είναι συζήτηση. Ίσως ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε και θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας πόσο χαίρομαι που τονίζετε ότι η εργασία μας είναι πραγματικά επικεντρωμένη στην ε, αξιολόγηση μεμονωμένων περιπτώσεων και ανηλίκων, διότι σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται μια συζήτηση μόνο επί ποσοτικού χαρακτήρα, πράγμα το οποίο είναι τελείως απαράδεκτο, διότι θίγει τα δικαιώματα του παιδιού και δημιουργεί δυσκολίες όταν εισέρχονται σε μια χώρα ή όταν αρχίζει η διαδικασία ενσωμάτωσης και καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει και είναι πάρα πολύ χρήσιμο να ανταλλάξουμε απόψεις για τις βέλτιστες πρακτικές διότι πάρα πολλά έχουν σχέση με την υλοποίηση, με την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας των ε, κανόνων που διαφέρουν ριζικά μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει βεβαίως να γίνονται σεβαστά τα υψηλότερα πρότυπα, τα υψηλότερα στάνταρ. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια αξιολόγηση επιμεμονωμένη ατομική βάσεω όσον αφορά την ηλικία, τη γενική κατάσταση του ανήλικα, τα ιατρικά θέματα, την... Ε, όλα, όλα τα χαρακτηριστικά που αφορούν την περίπτωσή του για να μπορούμε να εφαρμόσουμε τον καλύτερο τρόπο την νομοθεσία και τους κανόνες. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω έτσι για προσυζήτηση. Αν ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε για αυτό το θέμα είναι ένα νομοθετικό μέσον. Διότι ξέρω πόσο χρονοβόρα είναι η διαδικασία εισαγωγής και ενός νομοθετικού μέσου και συνεχεία μέχρι την εφαρμογή του. Το θέμα είναι πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε ένα τέτοιο εργαλείο, σε ένα τέτοιο μέσο ή να δούμε τι ακριβώς πράττουν τα κράτη-μέλη, το καθένα δηλαδή, για να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να βελτιώσουμε αυτές τις διαδικασίες για την καλύτερη προστασία των παιδιών. Σημαντικά βήματα λοιπόν, τα οποία θα ήθελα εγώ να υλοποιηθούν καταρχά. Εάν οπωσδήποτε θα ξεκινήσει μια νομοθετική διαδικασία, υπάρχει ο κίνδυνος τη οπισθοδρόμηση. Αντί του να προχωρήσουμε δηλαδή θα γυρίσουμε πίσω και γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε πού ακριβώς είναι τα προβλήματα, ε, τα θεσμικά, τα οποία εμποδίζουν μια θεσμική υλοποίηση των προγραμμάτων. Παραδείγματο χάρη είναι έλλειψη δυναμικού, έλλειψη φορέων, έλλειψη κατάρτισης. Ε, ίσως θα μπορούσαμε λοιπόν να εξετάσουμε το θέμα, όλα αυτά τα θέματα της εφαρμογής, τουλάχιστον να αναλύσουμε ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία αυτού του νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου. Ποια θα είναι Ελπίζω το Κοινοβούλιο με αυτή την έκθεση να συμβάλλει ε, δραστικά, αποτελεσματικά στην καλύτερη προστασία των παιδιών. Επίσης, Πρόεδρε, η συνεργασία με τρίτες χώρες, την οποία και εσείς αναφέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν γίνεται μία αξιολόγηση και κρίνεται ότι τα παιδιά αυτά ή ένας ανήλικας δεν χρειάζεται διεθνή προστασία όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων και άλλα προβλήματα. Είναι σημαντικό να αυξηθεί η συνεργασία στο, επίπεδο της Ένωσης για τον ε, επαναπατρισμό ή την επανένωση με την οικογένειά του. Πρέπει να συνεργαζόμαστε ε, καλύτερα με τα, τα, τους υπάρχοντες φορείς, τα, την υπάρχουσα υποδομή για να υπάρχει μια καλύτερη εγγύηση ότι τα παιδιά αυτά θα βρεθούν σε, μια, σε, μια, σε ένα ασφαλές πλαίσιο. Υπάρχει μια πρωτοβουλία στη Σουηδία που λέγεται ΕΚΟΝ για το Αφγανιστάν και το Ιράκ, όπου τουλάχιστον έχουμε διαπιστώσει τόση ότι βελτιώνεται η κατάσταση για συνόδευτους ανήλικες με καλύτερες ρήτρε ασφάλεια κλπ. που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλε περιπτώσει. Παρεπιπτόντως, με μεγάλη χαρά θα σας καλωσορίσω στη Σουηδία. τέλο Απριλίου η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών πηγαίνει στην Σουηδία και θα συζητήσουμε ακριβώς το θέμα αυτό και είσαστε προσκεκλημένοι. Ελπίζω να σας δω. Όπως και άλλες χώρες και η Σουηδία έχει προβλήματα και επιδιώκουμε την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Η κυρία Ζίμπελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς εδώ και αρκετές εβδομάδες γίνονται συζητήσεις σε πολλά σημεία για τα θεμελιώδη δικαιώματα, ε, τα, τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεμελιώδεις αξίες και βεβαίως μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συμπεριφορά μας έναντι ανηλίκων παιδιών, ε, φίβων, δεδομένου ότι αυτά τα προβλήματα παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και γι' αυτό ευχαριστώ ιδιαίτερα που συζητάμε και πάλι αυτό ε, το θέμα με την κυρία Γκρίμπεκ. Όμως ε, λείπουν συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό των ασυνόδευτων ανηλίκων αλλά και το πώς κατατάσσονται συνήθως βάσει ηλικιακής ομάδας και εν συνεχεία βεβαίως αποφασίζουν πώς θα γίνει η μεταχείρισή τους στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν βεβαίως και περιπτώσεις που κρίνονται ανάλογα με τις, ε, την κατάσταση του παιδιού, του ανήλικα. Ε, μερικές φορές ε, επίσης συνεργάζονται με μια οικογένεια. Υπάρχουν πολλές διαφορές στη μεταχείριση αυτών των <clears throat> παιδιών. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που παρατείναμε λίγο το χρόνο για τη διαβούλευση, γιατί μας λείπουν πάρα πολλές πληροφορίες και με, τον με την εισηγήτρια θα πρέπει να συζητήσω για να διευκρινίσω αυτές τις απορίες μου, αν μπορούμε δηλαδή να ξανασυζητήσουμε ορισμένα κρεμή ζητήματα και ε, τι ευθύνη έχουμε για την ε, μακρο, μακροχρόνια δηλαδή για το όλο θέμα. Ήδη Ξέρουμε, ελέγχθη, ότι ορισμένες προϋποθέσεις ήδη έχουν παγιωθεί ανεξάρτητα από την ε, έκθεση η οποία θα ψηφιστεί ή όχι. Δηλαδή υπάρχει ήδη ένα πακέτο το οποίο έχει αποφασιστεί, έχει εγκριθεί και μέσω αυτού μπορούμε να παρακολουθήσουμε κατά πόσο εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτού του υπάρχοντος ήδη πακέτου από τα κράτη-μέλη και να αναφέρουμε καλά παραδείγματα, διότι μέσα στο πλαίσιο το, της ανταλλαγής και της βέλτιστης πρακτικές μπορούμε να αναφέρουμε και τα καλά παραδείγματα. Ένα άλλο θέμα είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Συζητούμε σε πάρα πολλά σημεία και σε διαφορετικές επιτροπές τι πρέπει να γίνει, που ε, υπάρχουν ακόμα κενά και βεβαίως σε πολλές ε, σε πολλά σημεία χρειάζεται περισσότερο εντατική εργασία, όχι μόνο για την αγορά εργασία αλλά και για τους ανήλικες, τους εφήβους, τα παιδιά Ιδιαίτερα δηλαδή για τα άτομα αυτά, για τους πολίτες μας, για τους οποίους εκπονούμε όλη αυτή την πολιτική, πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα πώς χειριζόμαστε τον προϋπολογισμό. Θα ήθελα λοιπόν ε, να συζητήσω με τους συντηγητές περαιτέρω που έχουμε παγιωμένες ε, πολιτικές, που έχουμε ακόμα κενά και πώς μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να, να επιτύχουμε την καλύτερη προστασία των ανηλίκων. Ευχαριστώ. <clears throat> Κυρία Φλότρα. Σας ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Ναταλία Γκρίσπεκ για το έργο της. Νομίζω πραγματικά ε, μας δίνει μια βάση συζήτησης η οποία απεικονίζει πολύ καλά τα διακυβευόμενα και την κατάσταση στην Ευρώπη των ανηλίκων αυτών που είναι αφόρητοι. Αν φανταζόμασταν ότι ήταν τα δικά μας παιδιά στη θέση αυτών των ανηλίκων θα μας έπιανε φρίκι ότι οι πιο πολλοί από τους ανηλίκους είναι σε κατάσταση έγκλησης. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να γνωρίσουμε το ταχύτερο δυνατό την ταυτότητα και τις συνθήκες κράτησης αυτών των ανηλίκων και τα στοιχεία που μας δίνουν τα κράτη-μέλη είναι απόλυτα ανεπαρκή. Και όπως ελέγχθη, τα, οι ανήλικοι αυτοί είναι παιδιά. Πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν παιδιά πρώτα και σαν μετανάστες Δεύτερο, αυτό δεν είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εμφανίζεται στο σχέδιο δράσης της, γιατί βλέπετε ότι εκεί η προτεραιότητα δίδεται στην πρόληψη της έλευσης αυτών των ανηλίκων στην Ευρώπη και συγχρόνως στην επαναπρόθεσή τους στις χώρες προέλευσής τους. με τον τρόπο αυτό, με την ε, πολιτική αυτή αποτροπής της έλευσής τους και την εξασφάλιση της επιστροφής τους είναι οι προτεραιότητε της Κομισιόν, αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι η προτεραιότητα της δικής μας εργασίας. Αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει είναι να σκεφτούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό με τα νέα αυτά νομοθετικά μέτρα, με την ευρωπαϊκή στρατηγική, όπως θέλετε να την ονομάσετε, το ενοποιημένο πλαίσιο. Όλο αυτό Όλα αυτά είναι ερωτήματα ουσιαστικά τα οποία τα έθεσε και η κυρία Κοράτσα και η συγγήτρια. Είναι διαφορετικά τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλά ούτω ή άλλω θα πρέπει να δώσουμε το απαραίτητο ένδυμα σε αυτή τη ρύθμιση, ώστε η κατάσταση αυτών των ανηλίκων, που απεικονίστηκε σε πολλά ε, ευρωπαϊκά κείμενα, να μπορέσει να αντιμετωπιστεί με ένα ενιαίο τρόπο, με μία προσέγγιση για τους ανήλικες. Δηλαδή, ένα τρόπο αντιμετώπισης των μεμονωμένων, των ασυνόδευτων, ανηλίκων και όλα αυτά να μπορέσουν να συγκροτηθούν σε μια στρατηγική που να πλησιάζει παραδείγματος την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Ρωμά με την υποχρέωση να καταρτιστούν εθνικές στρατηγικές με σημεία αναφοράς σε κάθε κράτος μέλος Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να σκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο θα προωθήσουμε περαιτέρω αυτή την πρωτοβουλία που για μένα παίζει ένα κεφαλαιόδη ρόλο γιατί θα πρέπει να εξασφαλίσει την κινητοποίηση όλων των αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ασκήσει πίεση στις εθνικές αρχές για να μπορέσουν να τηρήσουν υποχρεώσεις που τους ανήκουν, δηλαδή να σεβαστούν το βέλτιστο συμφέρον αυτών των παιδιών και ανήλικων. στο <clears throat> πακέτο αυτό μέτρων υπάρχει και η οδηγία για την επαναπρόθεση. Σε αυτή την οδηγία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της μεμονωμένης εισόδου ανηλίκων ασυνόδευτων. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε αγαπητοί γείτονε, αλλά αν κάνετε λιγότερη φασαρία θα είναι καλύτερα. Ου, κύριε Παπα-Νικολάου, λέει ο πρόεδρος. Θα έπρεπε λοιπόν στα ευρωπαϊκά κείμενα να αναφέρεται μια προσέγγιση η οποία να μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω, να τύχει αξιολόγησης και να έχει ενοποιημένο χαρακτήρα για ένα κείμενο το οποίο θα αποτελεί την Ευρωπαϊκή Στρατηγική η οποία μετά θα εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη. Γιατί νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολο με άμεσο τρόπο να ρυθμίσουμε νομοθετικά όλα αυτά τα θέματα. Είναι Μεγαλό ο κίνδυνος ότι θα καθυστερήσει με τον τρόπο αυτό η βελτίωση της κατάστασης των ανηλίκων στην Ευρώπη. Και έχουμε επίση. Έχουμε πολλούς εταίρους, έχουμε τις κατευθυντήρες γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχουμε αναπτύξει εταιρικέ σχέσεις με αυτούς τους φορείς. Μπορούμε λοιπόν έτσι να βελτιστοποιήσουμε και τη χρήση των δημοσιονομικών πόρων, το αναφέρει και η συγγήτριά της για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το κοινωνικό ταμείο ή άλλα χρηματοδοτικά μέσα για να καλυφθεί η υποδοχή των ε, ανηλίκων και επομένως η, και η στέγασή τους, η εκπαίδευση και κατάρτισή τους, όλα αυτά που αναφέρονται. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν για μας πολύ χρήσιμο αλλά θα ήθελα να ξέρω και την άποψη της εισηγήτριας, γιατί συζητήσαμε το θέμα αυτό στην πρόσφατη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών. Αν θα ήταν σκόπιμο να έχουμε μία μελέτη για την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί εξ ονόματος του υπέρτερου συμφέροντος του πεδίου. Ποιε λοιπόν τέτοιε αποφάσεις θα μπορέσουν να αποτελέσουν ένα είδος προτύπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εδρεωθούν ως ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία των ανηλίκων. Δεν ξέρω τώρα αν αυτή η μελέτη έχει ξεκινήσει ή θα ξεκινήσει, αν έχουμε συμφωνήσει για αυτήν ή όχι. Ευχαριστώ λοιπόν την εισηγητρία. Ο κύριος Κέρκοφ. Κύριε Κύρκοφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι ενεπλάκησαν στη συζήτηση αυτή. Κρίμα που φεύγει η κυρία Κοράτσα Θα έκανε ένα σχόλιο για την πολύ θετική στάση που ακολούθησαν οι Σουηδικές Αρχές στην προετοιμασία της επίσκεψής μας τον Απρίλιο, όπου ελπίζω να μεταβώ και εγώ. Λαμβάνοντας βέβαια υπόψη το γεγονός ότι η Σουηδία θα υποδεχθεί την πολύ σημαντική διάσκεψη κορυφής του ΟΗΕ για την προστασία των, μάλλον, των παιδιών. Εγώ είχα παραστήσει αυτέ τι τις συνεδριάσεις δεκαετία του 90. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Κύριε Πρόεδρε, θέλω απλώ να σχολιάσω στο εξή ότι ενώ το έγγραφο εργασία παρουσιάζει τρει στόχου: ο πρώτο εστιάζει σε ένα ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο, αλλά εγώ το βλέπω να είναι το πιο ασθενές κομμάτι του εγγράφου. Τα άλλα δύο σημεία για τον τρόπο με τον οποίο οι ασυνόδευτοι ανήλικοι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι πολύ σημαντικό. Και εξίσου σημαντικό σ, είναι ο συνολικός στόχος του να αντιμετωπίσουμε το θέμα της λαθρεμπορίας ανθρώπων και της παράνομης μετανάστευσης. Γιατί αυτό φτάνει στην καρδιά των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Αλλά εδώ έχουμε μια δυσκολία. Είναι μια δυσκολία που έχουμε με όλε αυτέ τι συζητήσει που αφορούν τα παιδιά και του ανήλικου το θέμα του καθορισμού της ηλικία του ανηλίκου. Να μπορούμε να ξέρουμε αν κάποιος ή κάποια είναι πράγματι ανήλικος ή ανήλικη. Βέβαια στο έγγραφο εργασίας υπάρχει το τεκμήριο του ότι είναι ανήλικη. Δηλαδή τα επιχειρήματα τα οποία διατυπώνει το άτομο αυτό ή άλλη εξ του, καταρχήν θα πρέπει να θεωρείτε ότι είναι ισχυρά τα επιχειρήματα αυτά. Σε περίπτωση ε, αμφιβολίας θα πρέπει να είναι υπέρ του μαθητού ή καλύτερα υπέρ του ανήλικου σε αυτήν την περίπτωση ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί στους μηχανισμούς προστασίας. <clears throat> Νομίζω όμως ότι ο καθορισμός της ηλικία είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό, ίσως ακόμα πιο σημαντικό, είναι ότι ένας ασυνόδευτος ανήλικος, γενικά ένας ανήλικος δεν μένει για πάντα ανήλικος. Τι θα κάνουμε για να υπάρχει κάποια μεταβατική <clears throat> α, ρύθμιση για υποστήριξη αυτών των ατόμων όταν έρχεται κάποιος ως ανήλικος αλλά ενηλικιώνεται και κατά συνέπεια δεν καλύπτεται πια από αυτές τις ρυθμίσεις, αυτές τις πρόνοιες ως ανήλικος. Έχουμε κάποιο τρόπο ομαλής μετάβασης, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γι' αυτό λοιπόν <clears throat> με αυτές τις επιφυλάξεις που αναφέρω αυτές τις επιφυλάξεις θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Και επίσης, εγώ θα ήθελα να σας ε, ζητήσω να είμαστε πιο επιφυλακτικοί σε σχέση με την υπερβολική ρύθμιση. Το να έχουμε μια προσπάθεια να τα ρυθμίσουμε όλα μέχρι κεραίας, αυτό μπορεί να κάνει περισσότερο κακό, παρακαλώ. Αντίθετα, μπορούμε να δώσουμε την έμφαση στη συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών κτλ. μεταξύ αρμοδίων αρχών. Ούτω ή άλλω όμω όλα πρέπει να γίνουν για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα προστατεύει του ασυνόδευτου ανήλικε και θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα του προβλήματα. Ευχαριστώ. Κάποιο άλλο, ο κύριο Κλέη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω... Ε, στην έκθεση να δοθεί προσοχή στο θέμα του τράφικινγκ, της εμπορίας ανθρώπων και για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Ας μην είμαστε αφελείς. Υπάρχουν ολόκληροι κλάδοι δουλεμπόρων που με τρόπο κοινικότατο εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τη χάνουν υποδοχής έτσι ανθρώπινης και έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν μετά τα παιδιά αυτά πράγμα που οδηγεί ε, ενδεχομένως σε επόμενη μετανάστευση στα πλαίσια της συνένωσης των οικογενειών. Όταν μιλούμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα του παιδιού, θα πρέπει να σκεφτόμαστε και να τονίζουμε και την ευθύνη των γονέων. Διότι υπάρχουν γονείς που θελούσια στέλνουν τα παιδιά τους να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη για να πάρουν άδεια παραμονής και μετά να έρθουν και εκείνοι. δεν θα πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι επιβραβεύονται και όλες τέτοιες πρακτικές. Γιατί μακροχρόνια αυτή είναι η καλύτερη ε, μορφή υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ανηλίκων. Κάποιος είπε ότι θα πρέπει να συνεργαζόμαστε καλύτερα με τις χώρες προέλευσης και καταγωγής των μη, ε, συνοδευομένων ανηλίκων. Αυτά. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. and Madame Ευχαριστώ, κύριε Guillaume. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ την Αταλή Γκρισμπέκ για την έκθεση αυτή, την οποία θεωρώ πολύ θαραλέα, γιατί θέτει πραγματικά ξεκάθαρα τα ζητήματα. Και εγώ είμαι πολύ ευαίσθητη ε, για την ενοποίηση των διαφόρων κειμένων που ανέφεραν και οι άλλοι συνάδελφοι. Ε, εργάζομαι σε διάφορες εκθέσεις κι εγώ για το άσυλο και ε, είναι γεγονό αυτό. Μπορεί να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ε, ως προς τα αριθμητικά στοιχεία, τους αριθμού δηλαδή των ασυνοδευτών ανηλίκων στην Ευρώπη. Ε, θεωρούμε ότι το πρόβλημα του ασύλου για τους ανηλίκους είναι μάλλον δευτερεύον. Παραμένει όμως πρόβλημα και θα ήθελα να προσθέσω μερικά στοιχεία στη συζήτησή μας. Τα ζητήματα που αναφέρει η έκθεση είναι πάρα πολύ εύστοχα και αφορούν και πολλά θέματα του ασύλου, ας πούμε. Όχι μόνο τα διαδικαστικά. Και είδα στην έκθεση της Ναταλή Κρισπέκ κάποια σημεία σύγκλησης και θα πρέπει να τα προσέξουμε για να υπάρχει μια αντιστοιχία στον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα διάφορα προβλήματα και να είναι παρόμοιες οι προσεγγίσεις. Γιατί δεν συμβαίνει απαραίτητο αυτό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κράτηση. Οι ορισμοί που έχουν συμπεριφθεί στην οδηγία για την υποδοχή δεν συνάδουν με τα όσα προτείνει σήμερα η Ναταλή. Εν πάση να μην πω σε λεπτομέρειες, Δεν σας αναφέρω τα κεφάλαια με επικεφαλίδες για το πού χρειάζεται περισσότερο χτένισμα και συντονισμός. Το θέμα της υποδοχής των ασυνόδευτων ανηλίκων στην επικράτεια ε, της Ένωσης μπορεί να είναι προβληματικό. Γιατί διαφέρουν οι ορισμοί, οι προσεγγίσεις, θα πρέπει όλα αυτά να τα συντονίσουμε. Το θέμα της επιμέλειας. Η και Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα ορισμών. Ίσως θα πρέπει να το ελέγξουμε και αυτό ε, στο κεφάλαιο που έχει να κάνει ε, με τις απαιτήσει για την εκπαίδευση του κηδεμόνα, ε, την αποστολή του, τα καθήκοντα που αναλαμβάνει και εκεί χρειάζεται να ερμώνει στα κείμενα. Για τον καθορισμό της ηλικία έγινε μεγάλος λόγος. Βεβαίως στο θέμα του ασύλου ε, βλέπουμε ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ε, είναι προς το ενήλικες, είναι 16, 17, 18. Και ε, οι δοκιμές και οι έλεγχοι θα πρέπει να δούμε ε, ποιοι θα τις κάνουμε, με ποιο τρόπο, γιατί υπάρχουν και διζητικές μέθοδοι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις διάφορες διαδικασίες για τους ασυνόδευτους ανήλικους, και εκεί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, κοινά στοιχεία, να είναι μια κοινή προσέγγιση. Και το θέμα της κράτης που ανέφερα και πριν, προσωπικά και πολιτικά συμφωνώ απολύτως με τον ότι ο ορισμός με τον ορισμό μάλλον του ε, γράφου εργασία, ε, ότι ο σημερινό ορισμό δεν συνάδει με το διεθνέ δίκαιο και τα κείμενα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε έκτακτε όμω περιστάσει, εγκρίθηκε η κράτηση στην οδηγία για τις ε, συνθήκες κράτηση. Και εκεί λοιπόν χρειάζεται ενοποίηση των κειμένων για να είναι ισόρροπα και να ισχύουν παντού. Λοιπόν, η Κομισιόν τώρα έχει Α, έχει, θα έπρεπε να απαντήσει, να διευκρινίσει μια ερώτηση που τέθηκε από την κυρία Γκρίσμπεξ. Θέλει η Κομισιόν να λάβει το λόγο, διότι μετά θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για τελευταία φορά και μετά προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Η Κομισιόν. Ναι, πολύ σύντομα θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την ε, εισηγήτρια για την έκθεσή της η οποία περιέχει πάρα πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες και μια πολύ καλή ανάλυση του θέματος και ε, συμπληρώνει θαυμάσια το δικό μας πρόγραμμα δράσης επί το οποίο πέρσι το Σεπτέμβριο παρουσιάσαμε μια ενδιάμεση έκθεση, έκθεση μεσοπρόθεσμη οι ανήλικοι και οι είσοδό του στην επικράτεια δεν είναι καινούριο φαινόμενο στην επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολλούς λόγους, ε, ε, κακοποίηση στο σπίτι, στην οικογένεια, φτώχεια, ε, πολλοί λόγοι. Τώρα, γιατί τα παιδιά αυτά μετακινούνται και έρχονται στην επικράτειά μας, αυτό, ξέρουμε πολλούς λόγους, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να τα προσέξουμε, να τα φροντίσουμε και προστατεύσουμε. Γι' αυτό ακριβώς παρουσιάσουμε την έκθεσή μας. Ε, υπήρχε μια πολύ μεγάλη ε, κλίμακα, γκάμα αν θέλετε, πρακτικών που ε, επικεντρωνόταν στην μεταχείριση αυτών των παιδιών και γι' αυτό ακριβώς προσπαθήσαμε να συγκεράσουμε και να αναλύσουμε όλα αυτά τα μέτρα. Έτσι διαπιστώσαμε και περαιτέρω προβλήματα. Τα πολλά προβλήματα είναι εξαιρετικά τεχνικά. Παραδείγματο χάρη την αξιολόγηση κατά ηλικία, το θέμα της επανένωσης με τις, με τις οικογένειες. Είναι λοιπόν περίπλοκα και τεχνικά τα θέματα, αλλά υπάρχει περιθώριο συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και γι' αυτό έχουμε συστήσει και μία ειδική ομάδα, η οποία μία θα ασχοληθεί με την κυδαιμονία των παιδιών και η άλλη θα ασχοληθεί με το ζήτημα της επανένωσης, με τις οικογένειες. Επίσης, συνεργαζόμαστε με την Last η οποία ε, έχει περισσότερα στοιχεία όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή ε, και ε, συνεργαζόμαστε και με αυτή την οργάνωση, την EASO και θα συνεργαστούμε και για το θέμα της επανένωσης. Τώρα, στην νομοθετική πλευρά, λέει ο πρόεδρος, επίσης, Διακόπτει ο πρόεδρος. Παρακαλώ, ε, έρχονται τα μέλη μας μέσα στην αίθουσα για, την, ε, για να ψηφίσουμε, να αρχίσουμε τη διαδικασία. Παρακαλώ όμως να εισέρχεστε ήσυχα και να κάθεστε, διότι εκπρόσωπος της Κομισιόν μιλάει, έχει το λόγο. Επανέρχεται ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Λοιπόν, στο θέμα του νομοθετικού πλαισίου ε, έχουμε την οδηγία κατά της ανθρώπινης εμπορίας η οποία θετήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος δράσης και περιλαμβάνει συγκεκριμένα την προσέγγιση για το καλύτερο συμφέρον και προστασία του παιδιού θα πρέπει να αρχίσει η θέση ενισχύ αρχές αυτού του χρόνου και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή της στα κράτη-μέλη. Τα περισσότερα μέλη της ε, ΛΥΜΠΕ θα παρακολουθούν αυτή την κατάσταση, οι συζητήσεις συνεχίζονται και είναι περίπου και γι' αυτό η διαδικασία για τους ασυνάδευτου ε, ενήλικε ε, θα, βρίσκονται συνέχεια στο επίκεντρο, στην προτεραιότητα τη ατζέντα μα. Η, οδηγία επαν, επαναφοράς ε, ήδη έχει συζητηθεί και τώρα προσέχουμε ιδιαίτερα ορισμένε παραγράφους. Όσον αφορά τώρα τι γίνεται μετά τα 18 χρόνια, ε, μπορούμε να, να αναθεωρήσουμε ορισμένε διατάξει εφόσον δικαιολογείται και στους άνω των 18 ότι δεν μπορούν για συγκεκριμένους λόγους να ε, γυρίσουν πίσω στη χώρα τους. Και οπότε μπορεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να ληφθεί η απόφαση να μην ε, ε το παιδί. Ο, ο, ο, ενήλικας πλέον. Ο, ο πρόεδρος, πάλι διακόπτει ο πρόεδρος. Παρακαλώ, παρακαλώ. Συνάδελφοι. Παρακαλώ. Μην κάνετε τόση φασαρία. Ε, ε, βγείτε έξω από την αίθουσα αν θέλετε να μιλήσετε, όταν... αλλά μην κάνετε τόσο θόρυβο όταν μιλάει κάποιος στην αίθουσα. Λοιπόν, η Κομισιόν όσον αφορά την ε, εποπτεία του προγράμματος δράσης. Είπαμε ότι η τελική έκθεση θα παρουσιαστεί στο τέλος του 2014, αρχές 2015. Ο πρόεδρος, η κυρία Γκρίσμπαχ. Θέλετε να πείτε τίποτα, ε, να έχετε τον τελευταίο λόγο. Βεβαίως κύριε πρόεδρε, αλλά θα είμαι πολύ σύντομη. Γιατί κινδυνεύουμε να παρακάμψουμε τη συζήτηση εδώ, θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν την Κομισιόν για τις διευκρινήσεις που μας έχει δώσει. Πρέπει να είναι... <clears throat> Θα είναι δύσκολη η εργασία που έχουμε να κάνουμε και είναι απαραίτητο να έχουμε καλή συνεργασία με την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους και τους σκιώδεις συζητητέ και όλους τους άλλους οι οποίοι έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση αυτής της έκθεσης. Έχω λάβει υπόψη όλα αυτά που είπατε για την αντιστοιχία των ορισμών, για την ανάγκη συνεργασίας για την ε, ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών, ανταλλαγή πληροφοριών και στατιστικών. Το χιούμορ το οποίο χρησιμοποίησε ο κύριος Κίρκοφ για να θέσει το θέμα του πώς γιορτάσουμε τα 18 χρόνια ενός ανηλίκου και τι κάνουμε μετά. Όλα αυτά είναι κεντρικά θέματα τα οποία απαιτούν μια υπεύθυνη στάση από τη δική μας πλευρά. Υπενθυμίζω μονάχα κάτι που είπαν όλοι οι συνάδελφοι ανεξάρτητα από παράταξη σε σχέση με τη φύση του νομικού εργαλείου που θα πρέπει να προωθήσουμε. Εγώ προσωπικά διατύπωσα την άποψη ότι ίσως δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκρισταλώσουμε μια κάπως βαριά και επαχθή νομοθετική ρύθμιση που μπορεί να είναι αντιπαραγωγική. Αντίθετα όμως το να έχουμε μια στρατηγική ευρωπαϊκού χαρακτήρα για να αυξήσουμε και την συνειδητοποίηση και την αντίληψη του προβλήματος των ανηλίκων και την κατανόηση της ιδιαιτερότητός του θα ήταν πολύ χρήσιμο. Δεν είναι επειδή μερικές χώρες έχουν καλές πρακτικές και άλλες δεν έχουν καλές πρακτικές να αφήσουμε το θέμα αυτό να ρυθμιστεί μόνο από τα κράτη-μέλη. Η δική μας βάση ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και όλα τα άλλα κείμενα, όλα τα άλλα βασικά κείμενα τα οποία είναι και το υπόβαθρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι επειδή μερικά κράτη έχουν ή δεν έχουν κάποιες εθνικές ρυθμίσεις και δείχνουν ή δεν δείχνουν ενδιαφέρον για το πρόβλημα αυτό, να πούμε εμεί ότι δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε από κοινού. Αυτό θα πρέπει να το οδηγώ νήμα για μια κοινοτική, μια ενωσιακή καλύτερα προσέγγιση στο θέμα αυτό, ώστε να μπορέσουμε να προτείνουμε ρυθμίσεις οι οποίες να συγκλίνουν και οι οποίες να έχουν πάντα σαν γνώμονα το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού, ώστε ανεξάρτητα από το τι γίνεται ανεξάρτητα από την κατάσταση που λαμβάνει η χώρα, ένα παιδί είναι πάντα πιο ευάλωτο από ένα ενήλικα. Και ευχαριστώ να συνεχίσουμε την εργασία μας. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Και τώρα προχωράμε στην ψηφοφορία. Βλέπω ότι είναι πλήρες, ότι είναι πλήρης η αίθουσα με συναδέλφους οι οποίοι ήρθαν αδίμονες για την ψηφοφορία ή το καιρός. Δεν θα χρονοτριβήσουμε λοιπόν. Από ό,τι ξέρουμε, όπως ξέρετε όλοι μάλλον, από χθε αφαιρέθηκε ένα σημείο της ημερησίας διάταξης των ψηφοφοριών μετά από τη συμφωνία που κάναμε στην αρχή της πρωινής συνεδρίασης. Δεν θα, μιλήσουμε, δεν θα ψηφίσουμε λοιπόν την έκθεση Μακοβέ για το πάγωμα και την δίμευση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες. Πάμε στο πρώτο θέμα που είναι η πρόταση για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας με εισηγητή τον κύριο Μωράης. Αν είσαστε έτοιμοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ψήφι υπέρ του σχεδίου γνωμοδότησης του κύριου Μωράης. Κατά. αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το σύνολο της συστάσεως, ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. 39 3. υπέρ, 3 ψήφοι κατά, 6 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Μωράης, γίνεται δεκτή η γνωμοδότησή σας. Η κυρία Ινθρελ θέλει να κάνει μια δήλωση τώρα σε σχέση με το αποτέλεσμα αυτό της ψηφοφορίας. Εγώ κράτησα στάση αποχής, λέει ο κύριος Λουί Μισελ. Δεν είχα την κάρτα μου. Μία ακόμα αποχή, τέσσερις αποχές. Κυρία Ινφέλτ, θέλω να εκφράσω μία μειονοτική άποψη εξ ονόματος ομάδας μου. Κρατήσαμε στάση αποχής. Υποστηρίζουμε τους στόχους μεν τη πρόταση για διευκόλυνση προξενικών θεωρήσεων και υποστηρίζουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των ε, πολιτών της Ουκρανίας, οι οποίοι έχουν κάθε συμφέρον να αρθούν οι περιοριστικοί φραγμοί. Αλλά οι φιλελεύθεροι και οι δημοκράτες υποστηρίζουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και ανησυχούμε τα μάλα. Τα μάλα, ίσως και το ΕΛΚ να ανησυχεί, δεν είμαι σίγουρη. Ανησυχούμε πάρα πολύ για προτάσεις οι οποίες αφορούν μια νομοθεσία για τους ΛΟΑ, ΛΟΑ που επίκειται η ψήφισή τους στην Ουκρανία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι προαιρετικά, είναι ουσιαστικά. Γι' αυτό ζητούμε να αναβληθεί η ψηφοφορία. Ζητήσαμε να αναβληθεί η ψηφοφορία για να έχουμε περισσότερο χρόνο να εξετάσουμε το θέμα αυτό. Δεν το δέχτηκε η πλειοψηφία. Γι' αυτό η φιλελεύθερη ομάδα αποφάσισε να κρατήσει στάση αποχή. Εντάξει. Προχωρούμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία. Ο χάρτης Ευρωπαϊκή Ένωση πρότυπε διευθετήσει για την ελευθερία των μέσων ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Ρενάτε βέβαια. είναι πιο πολύπλοκο το θέμα αυτό. Έχουμε πολλές τροπολογίες. Ξεκινάμε. <clears throat> Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές απολύτω. 82. Θέλετε έλεγχο στην 81. έλεγχο για την 81. Άρχεται. Πέρας. 19 έναντι 27 απορρίπτεται πράγματι. Με τρεις αποχές. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά Αποχές. Δεκτή. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Έλεγχος για την 86. Άρχεται. Πέρας. 19 υπέρ, 27 κατά, μία αποχή απορρίφεται. 88 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 90 όχι, έχει, έχει εκπέσει. 95 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή Εκατό. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 106. Με προφορική τροποποίηση. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστή 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 1.19. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 120 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 123 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 127 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 133 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 138. Έλεγχο θέλετε για την 136. Μάλιστα. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 136. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 28 υπέρ 24 ε, κατά εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η συμβαστική 13 κατά αποχές εγκρίνεται 140 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα που πάμε στη συμβαστική όχι νομίζω ότι στην 142 υπάρχει ένα δεύτερο τμήμα που έχει διασωθεί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα θα περάσουμε στη συμβιβαστική υπαριθμό 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 141 έχει καταπέσει. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική υπέρθμο 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η συμβιβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 166 σε δύο τμήματα έτσι τμήμα πρώτον υπέρ Τα Αποχές. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. Αν θέλετε έλεγχο για το πρώτο, παρακαλώ. Επαλήθευση. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία για το πρώτο. Για την 166. Πέρασε. Ισοψηφία και μία αποχή. Οπότε... Τι ψηφίσατε? Υπέρ ή κατά. Γέοι νέοι που λένε και στην Αμερική. Άρα εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πηγαίνουμε στη συμβαστική 21 υπέρ. Ε, κατά αποχές εγκρίνεται. Η ε, συμβαστική 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 181 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 183 έχει αποσυρθεί. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 196 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 197 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 199 υπέρ. Κατά αποχές απορρίψεται. Τώρα έχουμε τις αιτιολογικές αναφορές και αιτιολογικές σκέψεις. Η τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η πέντε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, υπάρχουν μερικέ τώρα που καταπίπτουν και πάμε στη συμβιβαστική 26 26π, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 31 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 40 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 43 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 47 υπέρ κατά αποχές απορρίψεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 55 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ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 Λοιπόν, εδώ τι συμβαίνει. Θα τις ψηφίσουμε όλες μαζί, έτσι, ε, τις παραγράφους της νομοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού, με εξαίρεση τις παραγράφους 6 και 8. Λοιπόν, ψηφίζουμε πρώτα το σύνολο πλην των παραγράφων 6 και 8, έτσι. Ωραία. Υπέρ όλων των υπολείπων παραγράφων της νομοδότησης πλην ε, παραγράφων 6 και 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα η παράγραφη 6 και 8, υπέρ των παραγράφων 6 και 8. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται αυτές οι δύο παράγραφοι. Υπέρ της 8. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν και η 6 και 8. Και προχωρούμε στην ψήφιση του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Now closed. Ε, πέρας. Λοιπόν, να σας πω, είναι 47 υπέρ, 6 ε, κατά, χωρίς αποχές. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βέμπερ και συγχαρητήρια. Προχωρούμε τώρα στην επόμενη έκθεση. Παρακαλώ, ησυχία, προσέξτε με, παρακαλώ, ακούστε με. Ένα λεπτό, παρακαλώ, προσέξτε με, ακούστε τι λέω, γιατί έχουμε ακόμα δουλειά. Λοιπόν, τώρα θα ψηφίσουμε. Καλά. Voting now the report of... Θα ψηφίσουμε την έκθεση του κ. Παπα-Νικολάου για την απαλλαγή. Γενικός προπολογισμό τη Ευρωπαϊκής Ένωση. τμήμα 3, Επιτροπή, Απαλλαγή, ε, έτος, οικονομικό έτος 2011. Λοιπόν, είπαμε, τμήμα 3. Του κυρίου Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, καταρχάς, τροπολογία 1, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά τροπολογία 1 έκθεση κυρίου για την απαλλαγή. Ωραία. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. πέρα της ψηφοφορίας 19 υπέρ 30 κατά απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το κείμενο ως τροποποιηθέν. Ψηφίζουμε. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ και πάλι. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίας. 36 υπέρ Καμία ψήφος κατά 14 αποχές εγκρίνεται. Ωραία, προχωρούμε. Στο, τμήμα 9 της Εποπτικής Αρχής για την Προστασία Δεδομένων έχουμε μία τροπολογία. Ένα, ένα, υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ολόκληρο το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Ωραία. Δεκτή. 50 καμία ψήφος αρνητική, καμία αποχή ομόφωνα. Λοιπόν, σε μελιώδη δικαιώματα, οικονομικό έτος 2011 ή μάλλον η υπηρεσία σε μελιωδών δικαιωμάτων, το Ίδρυμα. Έχουμε τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίθηκε. 2 όχι καταπίπτη 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 ε, ε, αντικαταστάθηκε από μια προφορική τοπολογία της κυρίας Μάκοβεϊ. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 3. Άλλη μια προφορική τροπολογία της κυρίας Μάκοβέη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφο 3 με προφορική τροπολογία τη κυρία Μάκοβε, υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται, τροπολογία 7, υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται, τώρα ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. What do we have? Πάλι ομόφωνα με 50 ψήφους υπέρ. Ωραία. Τώρα θα ψηφίσουμε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας 2011. Απαλλαγή. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία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 Παράγραφος 5, προφορική τροπολογία του, της κυρίας Μάκοβε και της κυρίας Ματιού υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Όχι, τροπολογία, όχι. Τροπολογία 13, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το τοποποιημένο κείμενο, ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Αλλά άρχεται τώρα το σύστημα δουλεύει, πέρας ψηφοφορία. 46 υπέρ, καμία ψήφος ε, κατά, καμία απαλλαγή. Λοιπόν, ομοφωνία. Καμία αποχή, συγγνώμη. Τώρα και πάλι ο εισηγητή ο κ. Παπα-Νικολάου ψηφίζουμε την απαλλαγή τη Eurojust, τροπολογία 1, υπέρ. Κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 3, υπέρ. Κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. 4, υπέρ. Κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. 5, υπέρ. Κατά, αποχές, κατά, κατά. Λοιπόν, Ηλεκτρονικά για να είμαστε σίγουροι. Τροπολογία 5. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. 31 προς 16. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Ομοφωνία και πάλι 48 ψήφοι υπέρ. Έκθεση Παπα-Νικολάου για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Υπέρ, παρακαλώ, τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία. Or favor. Υπέρ κα, κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 καταπίπτει α είναι η τροπολογία 10 μάλιστα 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε το κείμενο ηλεκτρονικός έλεγχος πέρα της ψηφοφορίας πάλι ομόφωνα εγκρίθηκε με 47 ψήφους. Προχωρούμε. Απαλλαγή για την διαχείριση στα εξωτερικά σύνορα Frontex. Παράγραφος 1, ε, τροπολογία 1, ξεχωριστή ψηφοφορία της κυρίας Μάκοβεϊ. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος της τροπολογίας 2. Α, όχι. Του δεύτερου τμήματος της τροπολογίας 1. Του δεύτερου τμήματος. Ελέγχουμε. Παρακαλώ. Ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Έληξε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται, απορρίπτεται. 21 προς 25. Το δεύτερο τμήμα της πρώτης τροπολογίας απορρίφθηκε. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 3. Υπέρ. Αυτή την τροπολογία 3, ναι, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρα τη ψηφοφορία. 24 με 24, άρα απορρίπτεται. Εκτός αν κάποιος δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τώρα απορρίφθηκε. Τροπολογία 4, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται, 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, ψηφίζουμε την 5, παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Έληξε ψηφοφορία, έληξε, 48, ομόφωνα. Α, ψηφίσαμε ολόκληρο το κείμενο όπω τροποποιήθηκε. Συγγνώμη, έκανα λάθο. Και προχωρούμε στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία, απαλλαγή 2011, τροπολογία 1. Κατά, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. τροπολογία 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε όλο το κείμενο ηλεκτρονικά. Now closed. Έληξε ψηφοφορία. 48. Καμία αποχή. Α, και πάλι ομοφωνία. Προχωρούμε στην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 46 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, 0. Καμία αποχή. Ψηφίζουμε τώρα το σχέδιο γνωμοζώτησης με, σχε... με τη μορφή σχεδίου επιστολής από τον πρόεδρο σχετικά με τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων προϊόντα για τον άσπρο και την κατάργηση της οδηγίας 2001-20 ΕΚ. Μάλιστα. Α, ψηφίζουμε λοιπόν την, το, την επιστολή. Έγκριση σχεδίου επιστολής. Ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε. Τελείωσε. 48 υπέρ. Ομόφωνα. Εγκρίνεται. Και έχουμε μία ερώτηση για προφορική, μία απάντηση, μία προφορική, για εκ μέρους της Επιτροπής. Α, ερώτηση ε, για προφορική απάντηση. Μάλιστα. Ψηφίζουμε λοιπόν ε, την προφορική ερώτηση ηλεκτρονικά. Έληξε ψηφοφορία. Σαράντα τρία ψήφοι υπέρ τέσσερις κατά. Άρα λοιπόν η προφορική ερώτηση εγκρίθηκε και τώρα ολοκληρώσαμε, αν δεν κάνω λάθος, τις ψηφοφορίες. Σε ευχαριστώ, θα κάνουμε ένα σύντομα διάλειμμα πριν προχωρήσουμε ε, για So we wait or we ask. Why don't you ask them now before they leave the room? Okay. Hey. Oh, brother. Uh, excuse me, please. I had here in my order. Λοιπόν, Σύμφωνα ε, με την μερίσια διάταξη, το επόμενο σημείο, παρακαλώ ακούστε με. Σας είπα ότι θα κάνουμε ένα σύντομα διάλειμμα για να συζητήσουμε κάτι. So... Αλλά στην ημερήσια διάταξη έχουμε τους συντονιστές όπως ξέρετε. Παρακαλώ λοιπόν οι συντονιστές να μείνουν στην αίθουσα. Όσοι ψηφίσανε και δεν χρειάζεται να παραμείνουν, ε, να φύγουν παρακαλώ ήσυχα, να αποχωρήσουν ησύχως. Ε... Πιστεύω, λέει η ομιλήτρια, ότι υπάρχει μεγάλη βαβούρα στην Επιτροπή και υπάρχει σύγχυση και ένα μπέρδεμα και σήμερα στις ψηφοφορίες και χτες όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της ατζέντα, όσον αφορά την διανομή των καταλόγων ψηφοφορίας διότι υπήρχαν ε, πολλές συμβιβαστικέ τροπολογίες. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να συμμαζευτούμε σε αυτή την Επιτροπή διότι έχουμε, ε, δίνουμε την ακόνα έτσι λίγο ότι είμαστε διαλυμένοι, μια κακή εικόνα. Δεν λέω ότι είμαστε τέλειοι, κανένας δεν είναι τέλειος ε, και νομίζω ότι χρειάζεται μία βελτίωση. Take note. Of course you, you made your statement. Μία βελτίωση των εργασιών μας. Ο πρόεδρος βεβαίως σημείωσε την παρατήρησή σας. Αλλά όταν γίνονται προφορικέ ε, τροπολογίε που βάλλονται προφορικά ερωτήσει, δεν μπορούμε από νομική απόψεω να κάνουμε τίποτα να εμποδίσουμε αυτό το φαινόμενο.